Μετά από την ε, διακοπή των εργασιών το Δεκέμβριο μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου και βάση του άρθρου 7, ε, βάση του κανονισμού 78, θα δημοσιευθούν ε, τα πρακτικά, στα πρακτικά αυτά, οι νομοθετικές αυτές πράξεις. Για την Τετάρτη ζήτησε η παράταξη των Πρασίνων μία δήλωση της Αντιπροέδρου της, ε, ε, της ΥΠΑ εκπροσώπου για την Αλγερία. Η κυρία Χαουτάλα έχει το λόγο για να το αιτιολογήσει. Πρόεδρο, όπως αναφέρατε, η ομάδα μας προτείνει να, να γίνει δήλωση από την ύπατη εκπρόσωπο κατά προτίμηση με ψήφισμα για τα σε απίστευτες φρικαλαιότητες που έχουν ε, διαπραχθεί από την ομάδα Ισλαμιστών Μποκοχαράμ στη Βόρεια Νιγηρία. Μια ολόκληρη πόλη με 2.000 ανθρώπους φαίνεται να εξαλείφθηκε από προσώπου γης. Φαίνεται να είναι η πιο εκταμένη και φρικτή ε, ε, πράξη στην οποία έχει προβεί μέχρι στιγμής αυτή η ομάδα. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν να μπει αυτό το θέμα και η δήλωση στην ημερήσια διάταξη για την Τετάρτη υπέρ της ε, πρότασης ο κύριος Γκερέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μου θα θέλει να ε, υποστηρίξει ότι, λέγοντας ότι υπάρχει αυτή η δήλωση εκ μέρους της Αντιπροσώπου και θα προχωρήσουμε σε μια συζήτηση για αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί κατά επανάληψη στην Νιγερία και τα οποία πλέκτουν τη ζωή πολλών προσώπων και ιδιαίτερο στις ε, γυναίκες. Και, εν πάση περιπτώσει, θα προτιμούσαμε το ψήφισμα να εγκριθεί στην προσεχή συνεδρία της Ολομέλειας, γιατί θα συζητήσουμε ε, στο τέλος αυτής της εβδομάδας και δεν θα έχουμε πολύ χρόνο να το προετοιμάσουμε. Ναι, στη συζήτηση, ναι, στη δήλωση. Ε, ναι, βεβαίω θεωρούμε σημαντικό να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα και θα προτιμούσαμε η το ψήφισμα να εγκριθεί το Φεβρουάριο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με την πρόταση του κυρίου Γκερέρο καταρχήν να ακούσουμε μία δήλωση και στη συνέχεια να προβούμε στο ψήφισμα στην προσεχή συνεδρία. Okay. Ναι, νομίζω ότι είναι καλό το ψήφισμα και είναι ο καθήκον μας να το συζητήσουμε. Όποιο είναι υπέρ παρακαλώ να σηκώσει το χέρι. Κατά, αποχές, τότε το αποφασίζουμε, το ψήφισμα θα γίνει στην προσεχή συνεδρίαση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να μιλήσω κατά, αλλά απλά να ρωτήσω αν θα γίνει μια τόσο σημαντική συζήτηση την Τετάρτη ή μήπως γίνει την Πέμπτη το πρωί, όπου περισσότεροι ευρωβουλευτέ θα μπορούν να συμμετέχουν παρά να γίνει η συζήτηση αργά το βράδυ τη Τετάρτη, επειδή φαίνεται να μην χωράει κάπου αλλού αυτή η συζήτηση. Η πρότασή μου είναι δηλαδή να γίνει ναι, μεν η συζήτηση, αλλά την Πέμπτη το πρωί. Äh, ναι, δεν έχει γίνει ψηφοφορία και η κυρία Μουγκερίνη θα βρίσκεται εδώ όλη την Τετάρτη. Γι' αυτό έχει ένα νόημα να ακούσουμε τη δήλωσή τη, τη δήλωση είπα της εκπροσώπου Τετάρτη. Θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν ω τον περισσότεροι συνέδελφοι. Για την Πέμπτη δεν ε, υπάρχουν ε, αλλαγέ, αλλά θα ήθελα να σα καλέσω να παραμείνετε στι θέσει σα. Κυρίε και κύριοι,